ανάπτυξη, το διάλογο που θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Ψηφοφορίες παρακαλώ. Πρώτα έχουμε το κοινό ψήφισμα για το Ιράκ υπαριθμών δύο τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κύριε Ντεκιαζέ Πρόεδρε ο κύριος Μάουρο παρακαλώ να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με την τροπολογία του. Eh, ναι, ευχαριστώ. Να το διευκρινίσω. Δεν έχω στόχο να πω ότι οι χριστιανοί είναι περισσότερο μειονότητα από άλλες. Ωστόσο, είναι αλήθεια πως αυτήν την φάσεις της συζήτηση για το Ιράκ υπάρχει επιτάπητο η πρόταση να συγκεντρωθούν όλοι οι χριστιανοί σε μια μόνο ε, επαρχία. Αυτό είναι παράδεκτο. Γιατί όλοι όσοι είναι από τη Μοσούλ, το Κυρκούκ, ε, την Βαγδάτη να πάνε να εκτοπιστούν σε αυτό το γκέτο. Γι' αυτό και ζητάμε αυτή τη διευκρίνηση και αυτή θα το ε, μεταφέρουμε και στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών. Ευχαριστώ για την εξήγηση. Υπαριθμόν 3 τροπολογία υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κοινό ψήφισμα, κοινή πρόταση ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Το σημειώνω κυρία Τεκεζέρ. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Θιβέτ. Κοινή πρόταση ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και εν τέλει. Βυρμανία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τα πρακτικά της παρουσυνεδρίας θα υποβληθούν για έγκριση στο σώμα στην αρχή της προσεχούς περίοδου συνόδου, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μαζί με τα ψηφίσματα που ε, υιοθετήθηκαν σήμερα. Θα καταθέσω και τα ονόματα των όσων επισημένονται μέσα στα κείμενα. Ολοκληρώνεται έτσι αυτή